σε αυτή την ε, διεξοδική συζήτηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είναι κοντά μας δύο πολύ θαραλέοι αμύντορες ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Αζερβαϊτζάν. Η Λέλα και ο Άριφ Γιούνος ε, που συνοδεύονται από την κόρη του στην Άρα η οποία είναι εκείνη που έκανε πάρα πολλά για να φεθούν οι γονείς της ελεύθεροι. Φαντάζομαι, ε, συμφωνείτε μαζί μου κυρίες και κύριοι, πρέπει να τους χαιρετήσουμε θερμά. Θα θυμάστε όλοι ότι το 2014 η Λέλα Γιούνος ε, προτάθηκε για το βραβείο Ζαχάροφ ε, και εμείς ανησυχούσαμε τότε πάρα πολύ για την υγεία της ε, διότι ήταν κρατούμενη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ό,τι μπορούσε για να την αφήσουν ελεύθερη οι αρχές στο Αζερβαϊτζάν και από ό,τι βλέπετε τα καταφέραμε. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά και τιμή για μας μετά αυτό τον γολγοθά τράβηξαν, το να μπορούμε να τους δεχτούμε εδώ, να τους τιμήσουμε. Λέιλα, Γιούνος, Νάιρα, ευχόμαστε σε όλους σας υγεία, ευτυχία, τα καλύτερα για τη ζωή σας και να ξέρετε ότι και στο μέλλον θα σας στηρίζουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αγώνα σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ που μας επισκεφτήκατε. Η κυρία Μογκερίνη έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους αγαπητούς μας φίλους